Now we are ready. Dear friends, let me open, let me open the each... Λοιπόν, συνεδρίες Επιτροπής Ήτρε. Ο κ. Πολ Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τώρα έχω την κάρτα μου. Δεν είχα την κάρτα μου, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Α, ωραία. Ο, είδες, ήταν καλά, περιμέναμε λίγα λεπτά. Αν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο, θεωρείται εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Ουδέν σχόλιον. Δεν έχω κάποια ανακοινούση. Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης. 19 Φεβρουαρίου 2019. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδριάσης θεωρούνται εγκεκριμένα. ηλεκτρονική ψηφοφορία, σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια δοκιμή, δοκιμαστική ψηφοφορία, η οποία ξεκινάει τώρα, δοκιμή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ, όλα λειτουργούν καλά. Ας προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα. Σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως. Τροποποίηση του κανονισμού και ανάκληση 10 νομοθετικών πράξεων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων. Γιάννος Λεβαντόφσκι είναι ο εισηγητής. Αυτή η ψηφοφορία αφορά το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου Στη δεύτερη του Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία. Στη δεύτερη Ολομέλεια. Οπότε πάμε ψηφοφορία. Λοιπόν, στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων. Ονομαστική ψηφοφορία που αφορά την πρόταση, την προσωρινή συμφωνία που επετέφθη σε άτυπους τιμές διαλόγους. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Είναι εδώ ο εισηγητή. Όχι ακόμα, αλλά πιθανότατα σε μερικά λεπτά. Σημείο 5. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα δημιουργία του. Κ. Κασνοντεύσκη αφορά μερική συμφωνία επετεύθη με τη Ρουμανική Προεδρία στον τρίτο τριμερή διάλογο στις 19 Φεβρουαρίου 2019. Ξεκινάμε την ψηφοφορία Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Ο κ. Καζνοντεύσκη είναι ο συγκητής μας. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει για τη μερική συμφωνία που επετεύθη σε άτυπο τριμερή διάλογο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ευχαριστώ. Ξεκάθαρη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο το 6. Η δημιουργία του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Μασιμιλιάνο Σαλίνη, εισηγητής μας. Δεύτερος τιμερής διάλογος έλαβε χώρα 26 Φεβρουαρίου του 2019 που κατέληξε αποτέλεσμα και 13 Μαρτίου στην Κορεπέρ δόθηκε η τελική έγκριση αφού έγιναν κάποιες ευκαινήσεις για τα άρθρα 28 και 30. Στην Σύνοδο του Απριλίου, στη δεύτερη Σύνοδο του Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε μερική Συμφωνία που επετεύχθη σε άτυπο τριμερή διάλογο για το διαστημικό πρόγραμμα, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές. Συγχαρητήρια. Και πάμε στο σημείο 7. Δημιουργία του προγράμματος για την ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2000 το 2027. Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2019 καταλήξει συμφωνία. Θα ξεκινήσουμε με, τον, με την εισηγήτρια την κυρία Αντζέλικα Νίμπλερ. Μερική συμφωνία που επετέχθη στον άτυπο τριμερή διάλογο Ψηφιακή Ευρώπη, το σχετικό πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα. Υπέροχο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλους συγητέ, σκιώδεις συγητέ, Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί μου φίλοι, πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που δημιουργεί τον Ορίζοντα Ευρώπη, πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και ενοτομία που και καθορίζονται οι κανόνες για συμμετοχή και διάδοση του προγράμματος. Ωραία. Να σας πω μερικά λόγια για το θέμα. Λίγα λόγια για την υπόθεση. Λοιπόν, προσωρινή συμφωνία για τον ορίζοντα Ευρώπη, Horizon Europe, επετέφθη την περασμένη εβδομάδα στον έκτο και τελικό τριμερή διάλογο. Και πρέπει να πούμε ότι τα καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το σημαντικότερο που έχουμε. Είναι περισσότερα χρήματα που θα θέλαμε για το πρόγραμμα πλαίσιο. 120 δισεκατομμύρια σε τιμές 2018. Είναι κάτι σημαντικό που έχουμε μπροστά μας, ακόμα και με την ύπαρξη της μερικής συμφωνίας. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι βασικές διατάξεις συμφωνίας για τον κανονισμό του ορίζοντα Ευρώπη αφορά τη διεύρυνση τη θεματικής έρευνας για να αντιμετωπιστεί τα αντιμετωπιστούν προκλήσεις και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεγαλύτερη, ενέργεια, κλίμα, κινητικότητα να ξεχωριστούν, να καλυφθεί το κενό της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κλίμα να μπει σε όλες τις πολιτικές και αξιολόγηση σωστή και διαδικασία υποβολή σε δύο στάδια από είναι δυνατόν, ταχεία διαδικασία για έρευνα και καινοτομία, απλούστευση και επιμερισμός του βάρους για τους δικαιούχους, μείωση του βάρους για τους δικαιούχους, δυνατότητα προσφυγής και αναθεώρησης και τέλος οι συνημοθέτες συμφώνησαν επί πολύ ε, στενής παρακολούθησης και διατάξεων περί και υποβολής αναφορών. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό στην αρχή ε, του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη και βέβαια δεν συμφωνήσαμε επί κάποιου συγκεκριμένου στοιχείου διότι είναι αδύνατο, το ξέρετε πολύ καλά, είναι εντό αγγυλών για το Συμβούλιο το ποσό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δόθηκαν από τους συναδέλφους Ντανίκα και Κρίστιαν Έλλερ. Ντανίκα και Κρίστιαν Έλλερ που δεν μπορούν να παρίστανται απόψε. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ο κύριος Ρούμπικ. Ε, για μας είναι πολύ σημαντικό ε, το γεγονός ότι επιτεύχθηκε μια συμφωνία και θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους ε, Νίκα και Έλαντ και όλους τους συνεισηγητές κλπ. Ε, πιστεύω ότι είναι ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα και ήταν ε, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα αυτής της ε, θητείας. Ευχαριστώ. Competence. Oh, sorry is working. competence center and the network of national coordination. Το δίκτυο ε, εθνικών κέντρων, ε, συντονισμού των εθνικών κέντρων. Έχω μια, μια ενημέρωση από την κυρία εισηγήτρια, η οποία μας είπε ότι η δεύτερη τριμερή συνάντηση έγινε στις 22 Μαρτίου και πετεύθη κάποια πρόοδος. Παρόλα αυτά υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με κάποια ουσιαστικά σημεία της πρότασης, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτή την εβδομάδα. Η ψηφοφορία είναι μεθαύριο. Ωραία λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε. Σας διαβεβαιώ. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία, τα θέματα τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε σε αυτή τη θητεία. Το πρόβλημα είναι ότι στο Συμβούλιο έχει αλλάξει η Προεδρία και δεν ε, γνωρίζουμε κατά πόσο θα είναι παρόν αύριο το Συμβούλιο στην τεχνική συνεδρίαση και ε, κατά πόσο, είναι και κατά πόσο συνεπώς θα είναι δυνατόν να ληφθεί μια απόφαση την Πέμπτη. Ε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλήσεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το Συμβούλιο όσον αφορά το προπολογισμό αυτό θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ενώ εμείς ε, βάζουμε την, δίνουμε την προτεραιότητα στην ε, Κομισιόν. Και ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει να περάσει από την Ολομέλεια. Ας το αφήσουμε λοιπόν την Πέμπτη στην ημερήσια διάταξη και να δούμε πόσο θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε Πολ. Είναι πολύ σημαντικό που είσαι παρόν εδώ, σκιώδης, συγκητής, γιατί είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις από τη δική σου πλευρά, αλλά δεν νομίζω ότι πάρεις αντάλλη σκιώδης. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρούμπιχ. Ε, θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο σε σχέση με το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Κυβερνοασφάλειας ε, βιομηχανικής και του ε, Κέντρου ε, Βιομηχανικής Έρευνας. Θα περάσουμε λοιπόν στα διάφορα. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Έχετε κάποια παρατήρηση αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή Ήτρε, όχι. Ε, η προσοχή μας ε, είναι την επόμενη εβδομάδα, τριμερή συνάντηση. Καταρχήν και την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Την 1η Απριλίου η 1η Απριλίου έχει ακυρωθεί. Τη Δευτέρα Απριλίου λοιπόν στις 9 το πρωί έως τις 12.30 την Τρίτη. Η Δευτέρα Απριλίου είναι Τρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας.